Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίστε, προσθέστε τη ζώνη ασφαλείας ε, και ας απογειωθούμε. Ο συνάδελφος ε, ε, Λόνι θέλει να ξεκινήσουμε αμέσως ευτυχώς έχουμε νέους κανόνες. Δεν προεδρεύει ο πρεσβύτερος, αλλά ο αρχαιότερος εν τη υπηρεσία. Εγώ είμαι αυτός. Ευχαριστώ τον κύριο Λαβία και την κυρία Μπιουτικόφερ που είναι εισηγητές και δίνω το λόγο στον εισηγητή. Η γνωμοδότηση που προτείνω στην Επιτροπή σας για την οποία καλώ και τον κύριο εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών να μας υποστηρίξει ακολουθεί αυτά που είχαμε πει εδώ στην Επιτροπή τα τελευταία χρόνια ως προς τις δημοσιονομικές μας παρατεραιότητες. Πρώτον, θέλουμε να εκφράσουμε σαφώς την πεποίθησή μας ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση σοβαρών προκλήσεων όπως η σπάνιση των πόρων και άλλες. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός της Ένωσης έχει δυνατότητες συνεργιστικές και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προσθέτει κάποια αξία η Ένωση στη ζωή των πολιτών. Τρίτον, οι χρηματοδοτήσει πρέπει να ενδυναμώνουν την εφαρμογή της στρατηγικής 2020. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. been... Στο παρελθόν δεν αντέδρασαν τα θεσμικά όργανα με συνέπεια ως προς την εφαρμογή της ίδιας μας της στρατηγικής. Τι νόημα έχει να διατυπώνουμε στρατηγική, εντυπωσιακή, αλλά να μην βάζουμε τα χρήματα όπου χρειάζονται. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Και ελπίζω Ε, χρηματοδότηση που προβλέπεται τώρα στο 1α τη θεωρώ ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουμε τις προτεραιότητες της Ένωσης. Αυτό είναι μια επίκριση που παρακαλώ τους συναδέλφους να τη δεχτούν. Τέταρτον, προγράμματα όπως το Horizon 2020 ή η διευκόλυνση Connecting Europe πρέπει να έχουν επαρκή και χρηματοδότηση για να οθήσουν το πρασίνισμα της οικονομίας ως αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερα τα στηρικτικά προγράμματα για τις ΜΜΕ, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως οι επενδύσεις στις αναπτυξιακές των δυνατότητες. Αυτό δεν το λέω στην γνωμοδότησή μου, αλλά θέλω να το πω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του κόσμου. Δεν νομίζω ότι αυτά που έχει προβλέψει το κόσμο αρκούν. Και αν υπολογίζω σωστά τι θέλουμε να χορηγηθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το κόσμο και το Horizon 2020 τότε σε ευρώ του 2014 φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε καν αύξηση για τις άμεσες επιχορηγήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σύγκριση με το πρόγραμμα πλαίσιο του 7. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι σωστό. και αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τα πειραματικά προγράμματα για την ΕΤΕ σε, με ισοδύναμα κριτήρια για αυτά που εφαρμόζονται από πέρυσι δηλαδή μείωση των πληρωμών να αποφευχθεί. Και τέλος, ξέρω ότι εδώ η ΕΔΙΘ διαφωνεί καθώς και ορισμένοι άλλοι, θα ήθελα την υποστήριξή σας στην αντίρρηση του σχεδίου της Ήτρε για τα κονδύλια που είχαν χορηγηθεί από το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Αυτό σας προτείνω η διορία κατάθεση τροπολογιών λίγη την Πέμπτη το μεσημέρι. Παρακαλώ λοιπόν να το σημειώσετε. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Λαβία ως Γενικός Εισηγητής για τον Προπολογισμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είναι γνωστό σε όλους, η διαδικασία για τον προϋπολογισμό ξεκίνησε με την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε στην Ολομέλεια ήταν να ορίσουμε με δικά βασικά σημεία. Ανάπτυξη και στο πλαίσιο και μέσα στον όρο ανάπτυξη εντάσσονται πολλά από αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς τώρα στην ομιλία σας. Και δεύτερο το θέμα της απασχόλησης και κυρίως η απασχόληση των νέων. Όπως όλοι γνωρίζετε, το 85% των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη από το 2002 στο 2010 είναι θέσεις ε, που δημιουργήθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν απόλυτα για να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται σε όλο ένα πιο ευρύτερες αγορές. Είναι σαφές, όπως εξάλλου το αναφέρατε, Ο προϋπολογισμός του οποίου εργαζόμαστε είναι ο προϋπολογισμός του 2013, ο τελευταίο των δημοσιονομικών προοπτικών. εκεί θα έχουμε την εκφόρτιση όλων των μεγαλύτερων πιστώσεων ή υποχρεώσεων διότι όλες αυτές οι πιστώσεις υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει στο παρελθόν θα πρέπει πλέον να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι μας το ανέφερε σαφέστατα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι πέρυσι είχαμε σημαντική ζήτηση 16 δισεκατομμυρίων πληρωμών τους τελευταίους μήνες της χρονιάς που δεν μπόρεσε να εκταμιεύσει η Κομισιόν, μόνο 5 δις κατάφερε να πληρώσει. 11 λοιπόν δις στον τίτλο 1α και 1β, δηλαδή πολιτική έρευνα, για την έρευνα και πολιτική συνοχής. Αυτές λοιπόν οι πιστώσεις πληρωμών μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του 2012 και αυτό διατρέχουμε τον κίνδυνο να καταστεί τεράστιο πρόβλημα για τον προϋπολογισμό του 2013 εάν τα κράτη-μέλη μέσα στη χρονιά δεν εκπονήσουν έναν κατάλληλο διορθωτικό προϋπολογισμό. Όπως όλοι σας γνωρίζετε, η Κομισιόν αύριο το πρωί θα παρουσιάσει τη δική της πρόταση προϋπολογισμού. Εμείς ζητήσαμε από την Κομισιόν να είναι και φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική. Δηλαδή θα πρέπει να έχει συνέστηση και συνείδηση ότι πρέπει να απαιτήσει από τα κράτη-μέλη τις πιστώσεις για να μπορέσουν, τις χρηματοδοτήσεις, συγγνώμη, για να μπορέσουν τα προγράμματα να λειτουργήσουν. Αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, σίγουρα θα πρέπει να επενδύσουμε επί ορισμένων προτεραιοτήτων. οι οποίες αφορούν σε πολλά από τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή σας. Εγώ, ξέροντας ότι ετοιμάζετε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σας, αποφάσισα να κάνω αυτό το γύρο των Επιτροπών και να σας ακούσω για να είμαι ενήμερος και να σας εκπροσωπήσω στην εντολή του Τριολόγου στις 10 Μαΐου όπου εκπροσωπώ την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πριν ολοκληρώνω, να ολοκληρώσω, θέλω να, να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτο, προτεραιότητες. Πολλές από τις επιτροπές μας ζητούν να προσθέσουμε κονδύλια σε ορισμένες γραμμές του, του προϋπολογισμού. Αλλά σπανίως όμως εκτιμούν τις αρνητικές προτεραιότητες. Σε μια φάση λιτότητας και κρίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν έχουμε προγράμματα λιγότερο χρήσιμα, τα οποία δεν έχουν δυνατότητα δαπανών και στην στρατηγική μας θα πρέπει να τα θεωρήσουμε δευτερεύοντα ή περιθωριακά. Το να ζητάμε όλο ένα και περισσότερο είναι δύσκολο σε περίοδο κρίσης. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε γραμμές στον προϋπολογισμό που δεν αποτελούν προτεραιότητα. Δεύτερο, σχέδια πιλότη και οι προ... παρασκευαστικές δράσεις. Εμείς επ' αυτού έχουμε στήσει ένα χρονοδιάγραμμα έχουμε και το έχουμε ανακοινώσει στις διάφορες επιτροπές. Περιμένουμε από τις διάφορες επιτροπές τις προκαταρκτικές θέσεις, ε, ε, δράσεις συγγνώμη, και, τις, ε, και τα σχέδια πιλότο πριν από τις 10 Ιουνίου, ούτως ώστε η Επιτροπή Προϋπολογισμών να τα υποβάλει στην Κομισιόν και να έχει μία πρώτη αξιολόγηση μόνο τα σχέδια πιλότη που θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν θα χρηματοδοτούν. Θα χρηματοδοτηθούν. Τελευταίο. Αφορά στην επαναχρηματοδότηση του Ίτερ, έτσι όπως συμφωνήθηκε πέρυσι από τον Τρίλογο και τις δημοσιονομικές αρχές. Εμείς μέσα στα περιθώρια του τίτλου 1α είχαμε ένα περιθώριο επαναχρησιμοποίησης των 360 εκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά η αντιπαράθεση με το Συμβούλιο θα είναι ανοιχτή. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η δική σας προτεραιότητα για το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαβία για αυτή την εισαγωγή. Τώρα στη συνέχεια οι σκιώδεις εισηγητές των ομάδων. Καθένας τρία λεπτά προτείνω. Ο κύριος Ντάγκας παρακαλώ για το ΕΛΚ πρώτος. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά πρέπει να συμφωνήσουμε, θα λέγα, με την αξιολόγηση από πλευράς του εισηγητή και άλλοι, άλλα σχόλια ανέφεραν επίσης ότι το 2012 δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά, γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο προς μια νέα φάση σχεδιασμού. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες όμως. Και αυτό διότι η άποψη του εισηγητή είναι πολύ παρόμοια σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε πέρσι. Και γενικά, γενικά η πλειοψηφία των ιδεών αυτών είναι αποδεκτή και θα τις υποστηρίξουμε τις ιδέες και απόψεις αυτές. Όμως από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα όταν θα έχουμε το σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τελικά. Το σχέδιο αυτό του προϋπολογισμού μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες διαφορές απόψεων, όχι πολύ σημαντικές, αλλά παρόλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι Υπάρχει λόγος για να καταλήξουμε σε συνενετική θέση. Όμως το Ευρωκοινοβούλιο έχει ουσιαστικά στεναρή θέση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Συμβούλιο συνήθως όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού. Επίσης και μια άλλη δυνατότητα να εξετάσουμε να την δυνατότητα να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις για να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός. Ευχαριστώ για τη σύντομη γνωμοδότηση. Η κυρία Χέρτσοξ, στη συνέχεια σκιώδης εισηγήτρια, παρακαλώ έχετε τον λόγο για τους σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Μπιούτι Κόφερ. Και οι σκιώδης πέρυσι και φέτος συνεργάστηκαν καλά και βλέπω ότι τώρα έχουμε τους καρπούς της προσπάθειας αυτής. Βλέπω λοιπόν, ε, νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ακολούθησαν τη γραμμή <laughs> μας γιατί είναι πιο σημαντικό σε περιόδους κρίσεως να βρεθούν συνεργασίες και αλληλεγγύη μεταξύ χωρών μελών ως προς την, τα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης ε, που απορρέουν από το κεφάλαιο ανταγωνιστικότητας 1α. Δεχόμαστε λοιπόν την έκθεση του κυρίου Beauty Coffer μαζί με, με ορισμένες βέβαια. Να σας πω ποιες. Ένα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ε, στον προϋπολογισμό. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν πρέπει να αποκλείει από τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει μόνο η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών στον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα στο 1α, αλλά και μεταξύ των γενεών. Γιατί εμείς εξετάζουμε τη μικροχρόνια προοπτική. Είναι λοιπόν σημαντικό και αυτό το θέμα και θα θέλαμε να αναφέρεται στη γνωμοδότηση. Το σημείο 4 όμως μας είναι προβληματικό της γνωμοδότησης διότι δεν αφορά τον προϋπολογισμό του 13 αλλά για τα εργαλεία των δημοσιονομικών προοπτικών γενικότερα και δεν νομίζουμε ότι είναι κατάλληλος τόπος εκεί να μπει αυτό. Θα το τροπολογήσω μεν λοιπόν. Υποστηρίζουμε τα σχέδια, τα προγραμματικά σχέδια ομολόγων και μετά η Κομισιόν μας είπε ότι και ο Σκιώδης ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι ο τελευταίος χρόνος της προγραμματικής περίοδου και πρέπει να δούμε λοιπόν και τις πληρωμές όχι μόνο τις δεσμεύσεις. Και τέλος, για την ίτερ πρέπει να δούμε και τι έγινε την περασμένη εβδομάδα. Uh, Γιατί φαίνεται ότι δεν το κατάλαβαν όλοι. τα 100 εκατομμύρια από το 1α τεχνικά προήλθαν από το 1α αλλά τέθηκαν ως ένα εργαλείο ευελιξίας μέσα στο 1α δευτερεύον θέμα δηλαδή τεχνικό δεν είναι όμως από το FP7 το αναφέρει σαν FP7 στο 1α αλλά προέρχεται από το εργαλείο ευελιξίας. Αυτό να το ξέρουμε. Το άλλο θέμα που ρωτούμε την Κομισιόν είναι τα 360 εκατομμύρια που χρειάζονται για το 13 από πού θα προέλθουν. Η Επιτροπή μας νομίζω συμφωνεί ότι χρειαζόμαστε και άλλα χρήματα να μας διαθέσει το Συμβούλιο στα πλαίσια του εργαλείου ευελιξίας ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείου όχι μόνο για τα αποθέματα του FP7 αλλά και άλλων κεφαλαίων. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε η ΙΤΕΡ να έχει περικοπές ή να χρηματοδοτηθεί μόνο από το FP7. γιατί πρέπει όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους. Για το 2013 τίθεται λοιπόν το θέμα από πού θα προέλθουν τα 360 εκατομμύρια από την ευελιξία, από την έρευνα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι όμως μόνο από το FP7. Ευχαριστούμε κυρία Χέτσο. Ο, ο κύριος Ρούμπιχ ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Τον συνάδελφο Μπιουτικόφερ θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά επειδή ακριβώς η δική του προσπάθεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη σωστή χρονική στιγμή γίνεται. Μέσω της κρίσης χρέους θα είναι αναγκαίο κάποτε να επιστραφούν τα χρέη, να αποσβεστούν και η εξόφληση είναι κάτι που απαιτεί δουλειά. Δεν το κάνουν οι χρηματικές αγορές αυτό. Η πραγματική οικονομία θα το κάνει. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σχετικά και γι' αυτό πιστεύω ότι το πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2013 θα πρέπει να επιμείνουμε εμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα κονδύλια συνολικά να τα εξαντλήσει για αυτές τις δράσεις και να επικεντρωθούμε στους νέους, στις νέες επιχειρήσεις επιχειρήσεις που ε, δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές και φυσικά και για τις γυναίκες κυρίως οι γυναίκες που ασχολούνται με επιχειρήσεις ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή είναι οι πιο κατάλληλες για να είναι επικεφαλής επιχειρήσεων και να ιδρύσουν επιχειρήσεις ως επικεφαλής των επιχειρήσεων να βρούμε μια δυνατότητα από τον προϋπολογισμό ώστε να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. <clears throat> Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης ελπίζω να έχουμε καλύτερα καταρτισμένες γυναίκες επιχειρηματίες. Η κατάρτιση προέρχεται κατά κανόνα από την πρακτική την ίδια και γι' αυτό το πρόγραμμα Έρασμος για νέους επιχειρηματίες που ξεκίνησε από την Επιτροπή Ήτρε και που όπου 3.000 νέες γυναίκες που ασχολούνται με επιχειρήσεις μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με διάφορους τομείς και απεστάλησαν για να αποκτήσουν πείρα μια σημαντική αύξηση του προγράμματος Έρασμος για τους νέους επιχειρηματίες βλέπαμε από χώρα σε χώρα τι γινόταν αυτή η παλαιά προσέγγιση μπορεί να υποστηριχθεί μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε ακριβώς μέσα σε μια οικονομική κρίση καλά κατατισμένους δημοσιογράφους και γι' αυτό το πρόγραμμα Schumann στην Φλωρεντία για την πολυμορφία των μέσων είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι ακριβώς τα νέα μέσα δημιουργούν νέες, μπορούν να δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις απασχόλησης. Πολυμορφία λοιπόν των μέσων στον τύπο και υποστήριξη της δημοκρατίας που μπορεί να απορρεύσει. Γι' αυτό θα ήμουν πραγματικά στεναρά υπέρ αυτό το, αυτό το ε, πιλωτικό σχέδιο να διευρυνθεί, να επεκταθεί και να υποστηριχθεί. Τελευταία παρατήρηση. Συμφωνώ με τη συνάδελφο σε σχέση με το πρόγραμμα ITER. Νομίζω και εδώ πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα προερχόταν από το 7ο πρόγραμμα για την έρευνα. Χρειαζόμαστε πλήρη πλήρη εξοπλισμό της, του 7ου προγράμματος. Το ΊΤΕΡ θα δώσει αποτελέσματα τα επόμενα 20 χρόνια. Δεν θα είναι όμως μια συνεισφορά για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της κρίσης. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε από το πλαίσιο για την έρευνα να αντληθούν κονδύλια για το ΙΤΕΡ. Θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο η ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη να βρίσκεται στο επίκεντρο και η αποτελεσματικότητα στην παραγωγή και στην χρήση να υποστηριχθεί σε ευρύτερα πλαίσια. Γι' αυτό έχουμε το 7ο πρόγραμμα για την έρευνα και νομίζω ότι η σημαντική υποστήριξη στην Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι αναγκαία γι' αυτό. Yeah, ναι, σας ευχαριστούμε κύριε Ρουμπίχ. Δεν ζητούν άλλοι τον λόγο. Η Επιτροπή δυστυχώς δεν εκπροσωπείται. Τώρα έχει ο κύριος Μπιουτικόφερ την ευκαιρία να κάνει τις τελικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μόνο κάποιες λίγες παρατηρήσεις. Καταρχήν σε αυτά που είπατε εσείς ε, κύριε Τσαουντάγκας από κοινού ήδη πέρυσι προβληματιστήκαμε να δούμε σε ποιο σημείο αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ενδεχόμενα και από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό θα θέλαμε να παρεκκλίνουμε. Και εσείς επισημάνατε και είπατε ότι εφέτος σίγουρα πάλι θα αυτό θα είναι θέμα της συζήτησής μας. Πιστεύω ότι πράγματι θα συμβεί αυτό. Δεύτερον, το θέμα το δικό σας κυρία Χέρτσοκ, το ερώτημά σας για το σημείο 4 αυτής της γνωμοδότησης. Το σημείο 4 λοιπόν, τι λέει. Αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα έχουμε τον κεντρικό ρόλο αυτών των μελλοντικών προγραμμάτων Horizon 2020, Horizon 2020 και COSME σε αυτά στοχεύσατε και είπατε δεν είναι ακόμα αντικείμενο του προϋπολογισμού για του χρόνου. Όμως, στο δεύτερο σημείο αυτού του 4, του εδαφίου 4, διατυπώνεται μια αρχή που ισχύει και για τον προϋπολογισμό <clears throat> και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει στη σημασία του. Ήθελα να το επισημάνω αυτό. Τρίτον, για το σημείο ίτερ να επανέλθω σε αυτό και να πω το εξής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ο κύριος Λεβαντόφσκι ήδη υπέβαλε προτάσεις πως τα 63 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν ακόμα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν των διαβουλεύσεων για τον προϋπολογισμό προτείνει ο Λεβαντόφσκι όχι το σύνολο των 63 εκατομμυρίων αλλά τα δύο τρίτα των 63 δηλαδή 42 εκατομμύρια ετών να χρηματοδοτηθούν από τον τομέα της έρευνας και να έχουμε και 150 εκατομμύρια ευρώ από τον τομέα ICT, έρευνα ICT. Αν έτσι συγκεκριμένα τα θέσουμε ενώπιόν μας αυτά, τότε καταδεικνύεται για άλλη μια φορά με σαφήνεια πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπαμε όλοι, από κοινού όλοι μας ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ανταποκριθούμε. Και μάλιστα νομίζω αισιόδοξο πολύ θα ήταν κύριε Ρούμπιχ όταν, θα όταν λέτε εσείς ότι το ΙΤΕΡ ίσως 20 χρόνια θα δώσει κάποια συνεισφορά. Σύμφωνα με την άποψη των ερευνητών θα είναι μια εμπορική έρευνα που για την οικονομική διαδικασία θα μπορούσε να συνεισφέρει το νωρίτερο 50 χρόνια, μετά από 50 χρόνια όμως. Δηλαδή τα κονδύλια του προγράμματος έρευνας για ε, θα έπρεπε να επικεντρωθούν αυτή τη στιγμή έχοντας υπόψη την προτεραιότητα του κυρίου Λαβία, βιώσιμη ανάπτυξη, sustainable growth και job creation, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εδώ νομίζω είναι κάτι που σε σχέση με τη συνένεση είναι σημαντικό και για τα πιλωτικά προγράμματα που αναφέρατε. Και αυτό θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω ως έναυσμα, να δραχθώ αυτού και να πω ότι τα πιλωτικά προγράμματα αν έχουν κάποιες τέτοιες προτάσεις ε, και απόψεις οι συνάδελφοι για τέτοια πιλωτικά προγράμματα, μέχρι τις 30 Μαΐου πρέπει να κατατεθούν, ώστε να ακολουθήσουν την τακτική κανονική διαδικασία για την οποία μίλησε ο κύριος Λαβία. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπιουτικόφερ. Να επισημάνω κάτι. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 26 Απριλίου, 12 το μεσημέρι ως ήθιστε. Ευχαριστώ τον κύριο Λαβία που συμμετείχε στη συνεδρίαση και ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο έτσι τη ημερήσιας διάταξης. Το επόμενο σημείο είναι η Συμφωνία Εμπορία για το Εμπόριο για την καταπολέμηση των προϊόντων απομίμησης ε, ε, ως άκτα η συγγήτρια η κυρία Άντες Ντότερ. Την χαιρετίζω και της δίνω αμέσω τον λόγο. Παρακαλώ κυρία Άντες Ντότερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που επέτρεψε αυτήν τη συζήτηση στην Επιτροπή. Θα Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές για τη συνεργασία τους. Ξέρετε ότι η Συμφωνία Άκτα δημιούργησε πολλές συζητήσεις και μεταξύ των πολιτών αλλά και μέσα στην Ένωση σχετικά με το μέλλον του Ιντερνετ. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ειδικέ ευθύνε. Κυρίως αν δούμε και την όλη διάσταση που έχει πάρει το κίνημα των πολιτών σχετικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις για την πλαστογραφία. Πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς αναφέραμε τις επιπτώσεις της διακίνησης των εμπορευμάτων μαϊμού αλλά και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τη μεριά τους ανέφεραν ότι υπάρχει μία νομική ανασφάλεια για τις ΜΜΕ και για την ψηφιακή αγορά. Σε πολλές χώρες καταφέραμε να συζητήσουμε για τη δυναμική όλων αυτό, όλης αυτής της κατάστασης της ενδιάμεσης αγοράς. Λάβαμε θέση για την ουδετερότητα του διαδικτύου και όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή πρόσβαση. Πρέπει να, οι πολίτες να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκολία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Από τις θέσεις που ακούσαμε από τους διάφορους πρωταγωνιστές όλης αυτής της υπόθεσης διαπιστώνουμε ότι το άκτα μπορεί να είναι ουδέτερο έναντι του ίντερνετ. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της προστασίας των πνευματικών δεδομένων, δικαιωμάτων, συγγνώμη, και της πρόσβασης στο ίντερνετ. Εγώ στη γνωμοδότησή μου έγραψα ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να ζητήσει αυτή η συμφωνία να υπάρξει, να ισχύσει, αλλά όχι έτσι. στην εσωτερική αγορά της Ένωσης δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις για την περισυλλογή στοιχείων και πολλοί έχουμε διαφορετικές ε, απόψεις για τα αποτελέσματα των προϊόντων μαϊμού και τις επιπτώσεις ε, στο διαδίκτυο. Πριν όμως έχουμε δεσμευτικά μέτρα πρέπει να έχουμε νομική ασφάλεια και de facto ασφάλεια για την ισχύ της συμφωνίας. Πολλές διεθνείς οργανώσεις από τώρα όπως το G8 ε, ξεκίνησαν, άρχισαν μάλλον, να επιμένουν ούτως ώστε αυτή η συμφωνία να προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη της τα άλλα δικαιώματα. Η άκτα δεν κάνει όμως κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο, ένα μοναδικό μοντέλο για όλες τις πτυχές του διαδικτύου και αυτό μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγικό όταν διαπιστώνουμε την ετερογένεια των διαφόρων πρωταγωνιστών στην αγορά του διαδικτύου. Υπάρχει κίνδυνος να εγκρίνουμε μία συμφωνία που να μην, είναι, που να μην καλύπτει όλες τις καταστάσεις και αυτό μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο η Επιτροπή Βιομηχανίας και το θεσμικό μας όργανο των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού θα πρέπει να λάβει θέση για την προστασία των άλλων δικαιωμάτων και την ψηφιακή αγορά και θα πρέπει να αποφασίσει μια νέα στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εναντί του άκτα. Ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα με υποστηρίξει σε αυτήν φιλοδοξία και αυτήν την προσέγγιση και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στο μέλλον. Και ίσως θα έχουμε νέα μέτρα για μια νέα συμφωνία που θα προβλέπει όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής αγοράς. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Άντερστότερ. Τώρα οι σκιώδεις εισηγητές στη συνέχεια. Εκπροσωπώντας τον κύριο Κασπάρη, η κυρία Δεκαστήλιο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Κασπάρη είναι ο σκιώδης συγητής, όχι εγώ, ο οποίος για διάφορους λόγους απουσιάζει, οπότε είμαι εγώ τώρα η εκπρόσωπος της ομάδας μου. Αλλά θα πω και τη γνώμη μου. Υπάρχει μία αφετηρία που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Εγγύηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Χωρίς αυτήν την εγγύηση η ανάπτυξη και οι δυνατότητες απασχόλησης ζημιώνονται. Αν δεν αναγνωρίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία γεννώνται από την καινοτομία ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ομάδων ή προσώπων που δημιούργησαν, δημιουργών, τότε πραγματικά διαλύουμε ξεπουλάμε την κοινωνία που βασίζεται στην γνώση και στην δημιουργία. Όλοι συμφωνούμε αλλά αυτή τη στιγμή συμφωνούμε θα πρέπει να πασχίσουμε ούτω ώστε όλα αυτά να καταστούν εφικτά. Αυτό το οποίο θέλει η Άκτα ε, είναι, είναι μια εμπορική συμφωνία. Και, πως είπε και η συγγήτρια, πρέπει να το δούμε με μια θετική προοπτική. Αλλά όχι όμως βέβαιη ακόμα το ΑΚΤΑ προβλέπει έναν μηχανισμό για μια κοινή διεθνή προσπάθεια για τις καλύτερες προδιαγραφές προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Το ΑΚΤΑ δεν πλήττει τα άτομα ως προς την ψηφιακή της πτυχή, γιατί το ΑΚΤΑ είναι πολύ πιο πολύπλευρο που και έχει πολλά πεδία που δεν δεσμεύονται με το διαδίκτυο. Δεν έχει σχέση εδώ τίποτα με τα ατομικά δικαιώματα και την πρόσβαση στο ίντερνετ. Όλες οι εγγύησεις για την πράιβαση και την ασφάλεια ε, διασφαλίζονται. Και δεν αλλάζει το άκτα τα ε, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα οποιασδήποτε χώρας δεν θα αλλάξει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου πολλές φορές επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν αντεμβήξεις μεταξύ του περιεχομένου του άκτα και των όσων υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινοτικό κεκτημένο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι το ΑΚΤΑ αποτελεί αναγκαιότητα. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι λείπουν ακόμη στοιχεία για να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Αν αυτό είναι το, θα είναι το συμπέρασμα της ΙΝΤΑ, θα έλεγα να, υπάρχει μια, να γίνει μια άμεση δήλωση της Κομισιόν από κοινού με τους άλλους υπογράφοντες του Άκτα και να το πει καθαρά και εξάστερα το, το άκτα ξεκινήσαμε να το διαπραγματευόμαστε το 2008 και φτάσαμε πια στο 2012. Αν αναβάλουμε, αναβάλουμε, αναβάλουμε αυτή τη δράση, Σίγουρα χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα των στατιστικών, αλλά μεταξύ του 2009 και του 2010 η παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πνευματικών δικαιωμάτων αυξήθηκαν κατά 40.000 μέσα σε δύο χρόνια. Χάσαμε 150 εκατομμύρια ευρώ. Η ομάδα μου είναι κατά της απόρριψης του άκτα. και θα θέλαμε να υπάρξει μία διευκρίνηση της Κομισιόν μαζί με τους άλλους προσυπογράφοντες τη συνθήκη, αλλά θα ήθελα να γίνει γρήγορα. Διότι η ευημερία των κοινωνιών δεν δέχεται αναβολές και οι ώρες δεν είναι για, για τα πανηγύρια. Πρέπει να έχουμε τις βάσεις ε, για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την βαθιά κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλδημοκράτες εκπροσωπώντας τον κύριο Ντεάντζελης η κυρία Κατρίν Καουφμάν και να πω ότι κάπως καθυστερήσαμε είμαι γνωστός ότι είμαι αυστηρός για την τήρηση χρόνου τρία λεπτά πάνω κάτω. Ευχαριστώ καθένας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος του Ντεάγγελης που δεν παρίσταται σήμερα και θα σας πω τι ήθελε να δηλώσει εδώ στην Επιτροπή μας το άκτα παγώνει τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τροποποιήσει τα, ισχύοντα περί πνευματικών δικαιωμάτων και θα ήταν ένα βήμα επαναχώρησης από, σε σύγκριση με την έκθεση του Κοινοβουλίου για το ΙΠΡΕΝΤ 2 του 2006. Εκτός αυτού λυπούμαστε γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και είναι πολύ ασαφής οι ορισμοί στη συμφωνία η έκθεση Τζιγκαρέτη για το iPad 2 ήταν μία πρόοδος ως προς την, τον ορισμό της ενίας της εμπορικής κλίμακας, αλλά τελικά καταλήγουμε σε υπαναχώρηση για όλα τα υπόλοιπα. Το άκτα λοιπόν στην πράξη παραβιάζει ναι. τους στόχους της προηγούμενης νομοθεσίας. Η έκθεση Τζιγκαρέτη τόνιζε αυτά που τόνιζε η έκθεση Τζιγκαρέτη τα οποία εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία του 2006 δηλαδή ότι η παραβίαση από ένα χρήστη του ίντερνετ των δικαιωμάτων άλλων χρηστών δεν συγκρίνεται με τη συστηματική παραβίαση που κάνουν οι εταιρείες, οι υπεράκτιες εταιρείες. Τώρα καταργείται τελείως στην πράξη από το ΆΚΤΑ. Η ομάδα μας λοιπόν αποφάσισε να υποστηρίξει την πρόταση απόρριψης του ΆΚΤΑ παρά την προσφυγή στο δικαστήριο. Πρόθεσή μας είναι να υποστηρίξουμε πλήρως την απόρριψη της άκτας και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να και μπορεί να γίνει χωρίς καθυστέρηση στις διαδικασίες που ισχύουν για την Επιτροπή ΙΝΤΑ που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Εμείς θα γνωμοδοτήσουμε, πρέπει να γνωμοδοτήσουμε μέσα στο πρώτο ήμιση του Μαΐου. Πιστεύουμε ότι η κυρία Άντες Ντότερ έχει μια ισορροπημένη γνωμοδότηση που συμβαδίζει με πολλά από αυτά που έχουμε πει στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα με την εισηγήτρια σας. Κατευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε. Τώρα να σας διαβάσω τον πίνακα αγορητών Θα ήθελα να προτείνω να ολοκληρώσουμε τον πίνακα αγορητών και οι αγορητές να είναι σύντομοι αυτοί που άκουσαν το όνομά τους. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ επίμαχο θέμα. Έχουμε όμως και άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πιέζει ο χρόνος. Πρώτος, ο κύριος Ντέρεκ παρακαλώ. E, Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Η Συμφωνία Άκτα αφορά τρία σημαντικά θέματα. Εμπορικά δικαιώματα. Κάνουμε λόγο για το trademark για το άρθρο για, που προβλέπει τι θα γίνεται με τους χρήστες ε, του διαδικτύου και για τα δικαιώματα των τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών να εκμεταλλεύονται τα έργα τους οικονομικά. Σε σχέση με το πρώτο και τρίτο θέμα δεν βλέπω να υπάρχουν προβλήματα. Όμως για το άρθρο 27 αυτό δημιουργεί σημαντικές αμφιβολίες, ιδιαίτερα στα εδάφια 1 έως 8 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 4 τι συμβαίνει εδώ. Αυτό αφορά την ταυτοποίηση, την ταυτότητα του, των χρηστών του διαδικτύου που παραβιάζουν δικαιώματα ιδιοκτησίας. Παραβίαση λοιπόν δικαιωμάτων όσον αφορά και προσωπικά δεδομένα. Επίσης στην παράγραφο 6 γίνεται λόγος για τον εξοπλισμό που χρειάζεται και χρησιμοποιείται για την παράκαμψη της ε, προστασίας αυτής. Επίσης, κάτι άλλο, το 2005 η Ευρωβουλή πέριψε την γνωμοδότηση, την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για κάποιες ε, εφευρέσεις ε, που θα έκαναν χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών εγκεφάλων. Αυτό σημαίνει ότι το software, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι αντικείμενο λοιπόν διπλωμάτων εύρεση τεχνίας. Και γι' αυτό ένας προγραμματιστής μπορεί να σχεδιάσει νέο λογισμικό, νέο software εξ ονόματος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης. Δεν μπορεί να απαγορευτεί κάτι τέτοιο, πιστεύω, και σε σχέση με το, την παράγραφο 6 του άρθρου 27 απαγορεύεται ρητά μια τέτοια δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν θα αντέβαινε την αρχή της καινοτομίας όσον αφορά το λογισμικό, το software. Και αν δεν υπάρχει προκαθορισμένο δικαίωμα δημιουργού, τότε τα δικαιώματα τα πνευματικά ανήκουν σε εκείνον που συνέταξε, που σχεδίασε αυτό το λογισμικό. Άρα, τούτον λεχθέντων έχει απόλυτο δίκαιο η εισηγήτρια όταν κάνει λόγο για τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα που ε, εμπλέκονται εδώ έχοντας υπόψη την σημασία, την σπουδαιότητα της καινοτομίας, η πρόοδος πρέπει να υπογραμμιστεί, διότι η άκτα αντιβαίνει την καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά την τεχνολογία της πληροφορίας. Σας ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Πρόεδρε και θα ήθελα να σας πω ότι για την παρουσίαση της γνωμοδότησης των σοσιαλδημοκρατών ουσιαστικά είμαστε κατά της συμφωνίας ΑΚΤΑ. Την απορρίπτουμε για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα ο τρόπος με τον οποίο επετεύχθη αυτή η συμφωνία. Χωρίς δημόσια ανοιχτή συζήτηση, χωρίς να γνωρίζουμε τι ε, βρισκόταν υπό εξέλιξη. Επίσης είναι μια συμφωνία που δεν συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές μεγάλες χώρες που θα έπρεπε να εντάσσονται σε αυτή τη συμφωνία. Και το πιο σημαντικό είναι και το θέμα της ουσίας του περιεχομένου αυτής της συμφωνίας. Είναι συμφωνία εμπορίου και δημιουργούμε συμφωνίες για το εμπόριο επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης. Σε αυτήν όμως τη συμφωνία το αντίτιμο είναι υπερβολικά υψηλό και γι' αυτό είμαστε εναντίον της συμφωνίας αυτής. Η κυρία Στότερ μας έδωσε ένα πολύ καλό επιχείρημα και παρουσίασε σημαντικά, εξαιρετικά επιχειρήματα. Από πλευράς των σοσιαλδημοκρατών ο Ντέιβιντ Μάρτιν από την ομάδα μας έκανε την ίδια δουλειά λέγοντας ουσιαστικά ότι Πρόκειται για μια πολύ ισχνή, πενιχρή, κακή ποιότητα συμφωνία. Χάνουμε περισσότερα από ό,τι θα κερδίζαμε. Και γι' αυτό πρέπει να πούμε όχι, να την ε, καταψηφίσουμε. Και για τον τρόπο με τον οποίο η νέα συμφωνία των, ε, κοινωνία των πληροφοριών αντιμετωπίζεται, όλα αυτά τα στοιχεία τι σημαίνουν. Δεν είναι σωστή αυτή η συμφωνία, είναι πολύ αρνητική και γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση τη κυρία Άντερ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρούμπιχ παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέλια Άντερς Ντότερ, διότι φυσικά η Άκτα είναι ένα οικουμενικό θέμα, παγκόσμιο ζήτημα και πρέπει να δούμε πώς η Ευρώπη και στην συνέπεια, σαν συνέπεια αυτού και η πολιτιστική, η πολιτισμική βιομηχανία στην Ευρώπη πώς θα μπορέσει να δράσει σε ένα διεθνές πλαίσιο, παγκόσμιο πλαίσιο. Και αντιμετωπίζουμε πολυάριθμα προβλήματα φυσικά, για τα οποία στο τέλος τέλος πρέπει να βρούμε και απαντήσεις. Η νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου διαπίστωσε ότι η άκτα σε σχέση με την νομική τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχουμε όμως μία ενιαία νομοθετική διάταξη στην Ευρώπη και γι' αυτό η συζήτηση που διεξάγεται γύρω από τα θέματα της ΑΚΤΑ είναι πολύ σημαντική. Έχουμε και αντικρώμενα συμφέροντα. Έχουμε όλο, όλη τη βιομηχανία, τους καλλιτέχνες, τον τομέα της αναψυχής και διασκέδασης πολλοί που με πολλή δυσκολία και μεγάλο κόπο έκαναν δουλειά και πρέπει φυσικά να βρεθεί και η ανταμοιβή για αυτή τη δουλειά τους. Ερώτημα, ποιος θα πληρώσει αυτό το περιεχόμενο. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια μεγάλη διαφημιστική βιομηχανία, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο έχουμε στα χρηματιστήρια δισεκατομμύρια που διακινούνται από πολλές μεγάλες επιχειρήσεις μέσω διαφημίσεων που αξιολογούν το περιεχόμενο για πράγματα που πολλές φορές δεν υπάρχει αντίτιμο για αυτά και δεν πληρώνονται. Και υπάρχει αντικρουόμενο συμφέρον εδώ, υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ποιος θα πληρώνει τα κόστη αυτά στο τέλος τέλος και από πλευρά του συναδέλφου Γκέρεκ αναφέρθηκε αυτό. Υπάρχει το λογισμικό software που αναπτύσσεται και όλα αυτά στο διεθνές πλαίσιο και οι διεθνείς δυνατότητες που διανοίγονται, επιπρόσθετα έχουμε τις υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες. Ποιος πληρώνει λοιπόν για τα καλώδια, την καλωδίωση που χρησιμοποιείται για αυτές, για αυτές τις διαβιβάσεις. Και υπάρχει και, και σκληρή, α, σκληρή αντίθεση και αντιμαχία που στο σβέρκο των καταναλωτών διεξάγεται. Και δεν θα πρέπει εδώ να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δούμε ότι πρόκειται για σκληρά οικονομικά συμφέροντα και αντιπαραθέσεις. Ποιος θα είναι εκείνος που θα πληρώσει τα θέματα ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς θα καλυφθεί αυτό τι θα γίνεται. Και γι' αυτό ζητώ την εμπλεκόμενη βιομηχανία, τους εκπροσώπους της, να υποβάλουν εναλλακτικές δυνατότητες και μεταξύ τους να συμφωνήσουν και να μην μετακυλήσουν στον νομοθέτη όλα αυτά τα θέματα και να αναμείνουν να δουν ποιες εξελίξεις θα ακολουθηθούν. Γι' αυτό η άκτα είναι μια θετική βάση θα έλεγα ώστε η ευρωπαϊκή πολιτισμική βιομηχανία και τα δικαιώματά μας να τα υπερασπιστούμε διεθνώς και οι άλλοι αυτούς τους κανόνες που υπάρχουν στην Ευρώπη να τους σέβονται και να συμμορφώνονται με αυτούς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διεξαγάγουμε μια σοβαρή συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο να δούμε τι πρέπει να γίνει με την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσουμε, να δώσουμε λύσεις στα επίμαχα θέματα και με την Επιτροπή Διεθνούς ε, Παγκοσμίου Εμπορίου σε στενή επαφή να βρούμε συνετές λύσεις, ε, λογικές λύσεις. Αυτό πρέπει βραχυπρόθεσμα να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Ρόιχ, έχετε τον λόγο. Μάλιστα, λειτουργεί. Εντάξει. Κάποιες λίγες σκέψεις θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Το ζήτημα είναι πολύ περίπλοκο βέβαια. Πρώτον με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι αυτή η συμφωνία άκτα έχει μεγάλη προϊστορία και στην Ευρωβουλή. Υπήρξαν αποφάσεις που ελήφθησαν. Ασκήσαμε επικρίσεις πρώτα. Υπήρξαν ε, διορθωτικές κινήσεις και το Κοινοβούλιο είπε είναι εντάξει τώρα, δεν είναι καλός η υπόθεση. Έχω δυσκολίες τώρα, λίγο αργότερα να πούμε α όχι δεν πάει το πράγμα καλά, παρότι στο παρελθόν είχαμε πει ότι πήγαινε καλά. Πρώτο θέμα το οποίο με προβληματίζει αυτό. Δεύτερο θέμα, όποιος συζητά με ανθρώπους που παράγουν προϊόντα πνευματικής παραγωγής και ιδιοκτησίας, μουσικούς, καλλιτέχνες, ρωτάνε πώς ξαφνικά διεξάγεται μια συζήτηση δημόσια που δεν διασφαλίζει και δεν εκτιμά τα προϊόντα τους και πώς αλλάζουμε άποψη ξαφνικά. Αυτό με καθιστά πραγματικά βέβαιο και μου δημιουργεί προβλήματα να έχουμε τέτοια επίμαχα θέματα που δημόσια συζητώνται για την άκτα, μεγάλες διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες σε σχέση με τους νέους μεγάλα ερωτηματικά και όλα αυτά μπορούμε να τα αγνοήσουμε λέγοντας ένα όχι στην άκτα αν υπάρχουν αμφιβολίες για την άκτα, αν υπάρχουν θέματα που πρέπει να αποσαφινιστούν τότε πρέπει να αποσαφινίσουμε αυτά τα επιμέρους θέματα αρχών και όχι να εξοβελήσουμε το ζήτημα συνολικά εφόσον υπάρχουν ανάγκες διορθωτικών κινήσεων να διορθώσουμε αυτό το οποίο δεν βαίνει καλώς. Συγκεκριμένα, τι δεν βαίνει καλώς και τι πρέπει να κάνουμε να δούμε. Ιδιαίτερα αυτά τα οποία ισχύουν στην Ευρώπη και για το διεθνές εμπόριο ισχύουν και πρέπει να ισχύουν. Ε, δεν το κατανοώ πώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και τελευταίο ερώτημα, αυτό το οποίο ξαφνικά είναι δεδομένο νομικό για μας, νομική τάξη πραγμάτων, να αμφισβητείτε ξαφνικά. Ευχαριστώ. Ο Τζόρνταν. Η κυρία mm. Τζόρνταν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση που έγινε αυτούς τους τελευταίους μήνες θα λέγα είναι μάλλον ιδεολογική συζήτηση. Γι' αυτό χαίρομαι ότι σήμερα έχουμε μια επί συζήτηση. Οι συνάδελφοι και ο κύριος Ρούμπι για παράδειγμα υπέβαλαν πολύ ε, ε, λογικά επιχειρήματα. Λυπούμε γιατί δεν διατυπώσαμε τα σωστά ερωτήματα για λογαριασμό μας. Τι χρειαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Πρέπει να προστατεύουμε ως Ευρωπαϊκή Κοινωνία τα πνευματικά δικαιώματα γιατί είμαστε μια δημιουργική και καινοτόμα κοινωνία. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίζουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας ε, για τους παραγωγούς και τα άτομα. Τα προϊόντα τα οποία θα διακινούνται πρέπει να είναι συμβατά με την ετικέτα τους, ε, με Πρέπει να είμαστε πιο καινοτόμοι στις πρωτοβουλίες μας και να προστατεύουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ιδιαίτερα η ελευθερία πρέπει να διασφαλίζεται και να κατοχυρώνεται όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς καμία εποπτεία των ατόμων ε, ή λογοκρισία των χρηστών. Η άκτα υλοποιεί κάποιους συγκεκριμένους στόχους, συμφωνώ με αυτό. Όμως διαμαρτυρίες γίνονται παντού στην, διεξάγονται παντού στην Ευρώπη και στη Σλοβενία. Φοβούνται οι πολίτες να μιλήσουν ανοιχτά και δημόσια για την άκτα με ένα θετικό, πλαισ... Ε, με ένα θετικό τόνο. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ε, φωνές, όμως το θέμα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός όταν τόσοι πολλοί διαμαρτύρονται κατά της άκτα. Εκείνοι που διαμαρτύρονται κατά της άκτα ζητούν να καταργηθεί η άκτα αμέσως. Δεν συμφωνώ με αυτό όμως το άλλο ζήτημα από την άλλη πλευρά είναι ότι πρέπει να έχουμε μια επιστημονική πραγματογνωμοσύνη από ένα ανεξάρτητο σώμα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το σώμα εκείνο το οποίο θα έπρεπε να διασφαλίσει αυτή την πραγματογνωμοσύνη. Λυπούμε για το ότι απόλυσε, απεμπόλησε αυτή την ευκαιρία το Ευρωκοινοβούλιο το ότι δεν ζητήθηκε δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει. Θα έπρεπε να ξαναδούμε, να ξαναεξετάσουμε την άκτα, να τονίσουμε τις θετικές της πτυχές και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις αρνητικές. Το άρθρο 27 δεν είναι το μόνο σημαντικό άρθρο και έχω και ένα ερώτημα σε σχέση με αυτό. Υπάρχει κάποια δυνατότητα που να απομένει για μας για να ξαναδιαπραγματευτούμε το ζήτημα του άρθρου 27. Μπορεί να εξευρεθεί μια λύση για το άρθρο 27 που θα είναι αποδεκτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπαδία Κουτσέτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Άντερ Σότερ για την έκθεσή ε, ε, της για ένα θέμα τόσο καυτό. Πρέπει να βρούμε μία γρήγορη λύση όπως το είπαμε και εδώ. Αλλά η ταχύτητα να μην βλάψει την καλή λύση, τη σωστή λύση. Επ' αυτού η θεωρώ ότι η έκθεση Τζιγκαρετή πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση και βοηθούσε. Το άκτα έτσι όπως έχει σήμερα δεν είναι η καλή λύση και η καινοτομία θα πρέπει να, αποτελεί το βασικό μας, να αποτελέσει το βασικό μας σύμμαχο για να βρούμε τη σωστή λύση για την βιομηχανία, για τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους χρήστες. Τελευταίο θέλω να ξεκαθαρίσω και να προσπαθήσω να αποφύγω δηλαδή ότι όταν ε, αναρωτιόμαστε γύρω από το άκτα μας λένε είμαστε υπέρ των καλλιτεχνών ή κατά των ε, καλλιτεχνών. Ε, δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο μπερδεμένα. Έχουμε καλλιτέχνες που είναι υπέρ του άκτα, καλλιτέχνες που είναι κατά του άκτα, όπως και βιομηχανίες που είναι υπέρ και άλλες κατά. Ας δούμε λοιπόν τι, είστε, τι είναι καλό, τι είναι κακό και ας προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Όμως το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά σε αυτά τα επίπεδα δεν μπορεί να διορθώσει τη συνθήκη, αλλά εκεί πλέον που έχουμε φτάσει, το κοινοβούλιο μπορεί να πει μόνο ναι ή όχι. Αλλά εκεί που έχουμε φτάσει, τουλάχιστον να συζητήσουμε. Ο κύριος Ότμαρκ. Σας ευχαριστώ. Και σας και την εισηγήτρια. Είναι σημαντικό νομίζω να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα και την ελευθερία του ίντερνετ. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Εκπλήσωμε όμως πάντοτε όταν η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θεωρείται ως αντίθεση προς την ελευθερία του ίντερνετ. Συνήθως για τα πνευματικά δικαιώματα δεν λέμε τέτοια πράγματα. Η Επιτροπή μας συχνά τόνιζε πόσο σημαντικά είναι πόσο σημαντική είναι μια συνεπής αντιμετώπιση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων για τις ευρεσιτεχνίες και για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς προς την καλύτερη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν βλέπουμε. Αυτό δεν το βλέπουμε συνήθως ως αντιφατικό με την ελευθερία της πληροφόρησης. Γιατί να διαφέρει το ίντερνετ από άλλα μέσα είτε θα προστατεύουμε την πνευματική ιδιοκτησία είτε όχι. Χρειάζονται ίσως βέβαια κάποιες προσαρμογές στην πραγματικότητα των νέων τεχνολογιών, αλλά πρέπει επίσης βασιζόμενο στις συμπεράσματα της νομικής υπηρεσίας και άλλες νομικές νομοδοτήσεις να πω ότι δεν υπάρχει εδώ καμία ασυνέπεια ούτε τίποτα φοβερά καινούριο στην άκτα. Εδώ φαίνεται κυνηγάμε φαντάσματα. Εγώ ποτέ δεν είδα να υπάρχει καμία πραγματική απειλή όπως λένε ορισμένοι. δεν πρόκειται για καμία παραβίαση της ελευθερίας του ίντερνετ. Ίσως όσοι αντιτίθενται στην άκτα δεν είναι υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Για μένα είναι απαραίτητο να είμαστε συλλογικοί. Άμα θέλουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να δεχτούμε και την άκουτα και ούτε οι νομικές υπηρεσίες βρήκαν κανένα ψεγάδι στην άκτα. Και παρόλο το σεβασμό που οφείλω στην εισηγήτρια δεν το βλέπω ούτε στην γνωμοδότησή της στην απόδειξη ότι παραβιάζεται η ελευθερία. Δώστε μας παραδείγματα. Ή αλλιώς πέστε μας ότι είστε κατά της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία όμως δεν παρεμποδίζουν την ελευθερία της πληροφόρησης. Το θέμα είναι αν τα θέλουμε ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ αυστηρός στην προάσπιση της ελευθερίας του ίντερνετ. Και βλέπω ότι η άκτα ήδη διόρθωσε ορισμένες από τις παλαιότερες διατάξεις της όπως την αυτόματη φραγή κτλ. Αλλά παρακαλώ δώστε μας συγκεκριμένα παραδείγματα παραβιάσεων όπως λέτε. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να διασφαλίσουμε, να καταλάβουμε αν πρόκειται για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή όχι. Ήμπλε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Άμεσα μπορώ να συνεχίσω αυτά που είπε ο συνάδελφος Εκμακ. Hunting a ghost, κυνηγώντα φαντάσματα. Αυτή την εντύπωση είχα και εγώ τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τον τρόπο που συζητήθηκε η Συμφωνία Άκτα τον τελευταίο καιρό. Έκανα τον κόπο να διαβάσω όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές την Άκτα. Και όλες αυτές οι εντάσεις και φορτισμένες αντιδράσεις είναι κάτι που δεν μπορώ να κατανοήσω και με την Νομική Επιτροπή όπως είπαμε έχουμε δώσει εντολή από την Νομική Επιτροπή που επιβεβαιώνει αυτά που πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν για άλλη μια φορά ότι υπό το ευρωπαϊκό πρίσμα δεν μπορεί να δει κανεί ότι η άκτα για την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας αλλάζει κάτι για η συμφωνία αυτή είναι μια enforcement συμφωνία υλικό δίκαιο, υλικό της σημερινής διεργασίας νομικής τάξης δεν ρυθμίζεται διαφορετικά. Όποιος πιστεύει κάτι διαφορετικό, το ανέφερε ο συνάδελφος Φεκμακ, να μας αναφέρει το εδάφιο, την παράγραφο, το παράθεμα σε αυτή τη συμφωνία όπου σε σχέση με το υλικό δίκαιο υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και όταν λέει κανείς να αλλάξει το πλαίσιο προστασίας ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο τότε σε σχέση με αυτές τις προτάσεις να διεξαγάγουμε τη συζήτηση Έχω ανοιχτό πνεύμα για τις, ε, τους φόβους και τις αμφιβολίες. Πρέπει να συζητηθούν σε βάθος τα θέματα και ίσως και να αλλάξει το πλαίσιο προστασίας ε, των δικαιωμάτων δημιουργού, πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Αλλά κατά τα άλλα δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να αρνηθούμε την έγκριση της άκτα. Εκατό φορές μπορούν να εξετάσουν οι νομικοί αν είναι συμβατό ή όχι το πλαίσιο αυτό. Θέλουμε να υπάρχει νομική βεβαιότητα, αλλά βασίζομαι σε αυτά τα οποία είπε η νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι φιέστατοι άνθρωποι, πολύ καλά εκπαιδευμένοι και μας υπέβαλαν αυτή τη σύσταση. Έτσι λοιπόν συμφωνώ, πρέπει να εγκρίνουμε την άκτα και όχι να την απορρίψουμε. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή παρακαλώ τώρα. Thank you, Madam um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας πω και εγώ μερικές σκέψεις γρήγορες. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Γιατί η άκτα δεν φλάπτει τους πολίτες αλλά βοηθάει τις εταιρείες, ιδίως τις εταιρείες που εξάγουν διεθνώς και που θίγουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας Mm. Είναι λοιπόν η άκτα απαραίτητη για να βοηθήσει την Ευρώπη στο εμπόριό της και την ανταγωνιστικότητά της. Κατά τις διαπραγματεύσεις προσέξαμε ιδιαίτερα να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην άκτα μάλιστα παραπάνω από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία και ενωσική νομοθεσία Επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων. Καμιά φορά το λέμε δύο και τρεις φορές το ίδιο άρθρο όπως το 27. Παρόλα αυτά παραμένουν αμφιβολίες όπως υπόθηκε και σήμερα. Αλλά είναι αμφιβολίες χωρίς παραδείγματα συγκεκριμένα. Λόγω των αμφιβολιών αυτών η Κομισιόν έστειλε την άκτα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παρέπεμψε. Μπορεί όπως ζήτησε και ο Επίτροπος και η Προεδρία να χρειαστεί να περιμένουμε την τελική άποψη για την νομιμότητα ή μη της άκτας που θα δοθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τότε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τη βεβαιότητα ότι έχουμε την τελευταία λέξη για αυτό το πολύπλοκο θέμα. Υπόθηκε πολλές, αναφέρθηκε πολλές φορές το άρθρο 27, το οποίο όμως δεν παρεμποδίζει καθόλου την ελευθερία του Ιντερουνέτ. Οι διατάξεις του είναι προαιρετικές, αναφέρει ορισμένες αρχές που ήδη εφαρμόζονται από υπάρχουσα νομοθεσία εδώ και 10-12 χρόνια και που δεν παρεμποδίζει την άνθηση του ίντερνετ δεν περιέχεται εδώ καμία απειλή για τον χρήστη και τη χρήστρια. Όσο για τις διαμαρτυρίες βλέπουμε ότι πολλοί από τους διαμαρτυρωμένους αναγκάζονται να παραμείνουν σε θέματα ορισμένων κανόνων του copyright. Αν απορριφθεί όμως η άκτα δεν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Η άκτα είναι κανονιστική πράξη. Το ότι θα χρειαστεί αναμονή για να βγει η απόφαση του δικαστηρίου δεν σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να περιμένει και την εξέταση άλλων σχετικών προτάσεων της Κομισιόν για τα πνευματικά δικαιώματα, για τις άδειε, για τις εβούρες ή τεχνίες κτλ. Η Κομισιόν λοιπόν και ο υπεύθυνο Επίτροπος θα ήθελα να πούν στο Κοινοβούλιο ότι ίσως θα έπρεπε μεν να περιμένει την τελική απόφαση του δικαστηρίου και να μην απορρίψει ήδη από τώρα κάτι που το υποστηρίζει τεράστιος αριθμός συνδικάτων, εταιριών και καλλιτεχνών και καλλιτεχνιδών. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ και, στην, και την Κομισιόν για την παρουσία της. Για μένα είναι ενθαρρυντικό να διαπιστώνω ότι η Επιτροπή μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τόσο δύσκολη συζήτηση ενιαία. Αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία. Πολλοί μίλησαν πόσο σημαντικό είναι για μας το σινεμά, η μουσική, αλλά το άκτα είναι κάτι το πολύ ευρύτερο Πολλά παίζονται με το άκτα για την ψηφιακή οικονομία. Και αναρωτιόμαστε αν το άκτα αποτελεί ένα μέσο για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο των απαραίτητων μέτρων. Μου φαίνεται φάνερο ότι στο μέλλον χρειαζόμαστε μια πιο διαρθρωμένη συζήτηση. Το άκτα δεν φαίνεται να είναι η καλύτερη πλατφόρμα για την ειδική συζήτηση των διαφόρων τομεακών συζητήσεων. Εγώ αναμένω τις τροπολογίες και μετά να δούμε ποια θα είναι η συζήτηση. Να σας πληροφορήσω για το χρονοδιάγραμμα. Εμείς ε, ζητήσαμε να έχουμε μία αναβολή. Θα έχουμε την απάντηση όμως αύριο. Εάν δεν υπάρξει αυτή η αναβολή για ένα μήνα στο χρονοδιάγραμμα, οι τροπολογίες θα έπρεπε να κατατεθούν στις 27 Απριλίου μόνο στα αγγλικά και θα ψηφίσουμε στις 8 Μαΐου. Αν τώρα αύριο η Ίντα μας ανακοινώσει ότι όντως δέχεται αυτήν την αναβολή, τότε θα σας στείλουμε ένα email, σε όλους φυσικά, οι τροπολογίες παραμένουν με προθεσμία την 27η Απριλίου, αλλά μπορούν να κατατεθούν σε όλες τις γλώσσες. Αλλά η ψηφοφορία θα γίνει στις 30-31 Μαΐου. Ξέρετε ότι στις 10.30 έχουμε κοινή συνεδρίαση με τις μεταφορές. Ας κάνουμε τώρα έναν αγώνα δρόμου για να δούμε αν καταφέρουμε να εξετάσουμε το τελευταίο σημείο του κυρίου Σιμάνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζετε η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία είναι ένα ευρύτερο εγχείρημα που θέλει να συνεισφέρει από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών προς, προς την Ανατολική Ευρώπη και προς τον Νότο να συγκλίνουν. Είναι πολιτικό εγχείρημα και έχουμε και ένα χρηματοδοτικό μέσο Όσον αφορά την ενέργεια, ενεργειακά θέματα που πρέπει να αποτελούν κύριο στοιχείο της πολιτικής γειτονίας, οι όμορες χώρες έχουν μεγάλο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν όσον αφορά την διαμετακόμιση, το διαμετακομιστικό εμπόριο και την παροχή φυσικού αερίου, πετρελαίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να διευκολυνθούν όλα αυτά πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα ισχύει στη διάθεσή μας και που πρέπει να συσχετίζεται με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, με τα πρωτόκολλα, με την χάρτα ενέργειας, ενεργειακών θεμάτων και πρέπει και να οδηγεί σε απελευθέρωση των αγορών μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει εδώ το τρίτο πακέτο η ασφάλεια η ενεργειακή είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Η πολυμορφοποίηση όσον αφορά αυτά τα προϊόντα και την παροχή τους, αυξημένος ανταγωνισμός, μείωση εκπομπών ρήπων, όλοι αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν λοιπόν. Και για αυτούς όλους τους λόγους υπέβαλα και την πρόταση αυτή για και τις τροπολογίες που έχουμε σε σχέση με αυτή την έκθεση από πλευράς της ε, κύριας της αρμόδιας επί της ουσίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Πιστεύω ότι με τις τροπολογίες αυτές θα καταφέρουμε στο τέλος να πετύχουμε ένα καλό κείμενο και μπορούμε αν είμαστε αρκετά γρήγοροι να έχουμε μια καλή πρόταση που υποβάλλεται στις διαδικασίες συναπόφασης με την ε, συμμετοχή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ γόνιμη καρποφόρα συνεργασία με αυτούς και με μια περαιτέρω συνάντηση που θα έχουμε με τους σκιώδης μπορούμε να πετύχουμε μια πολύ καλή πρόταση εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κόσμος αλλάζει και εξελίσσεται και χαίρομαι για την εφαρμογή αυτών των δημοσιονομικών πλαίσιων ε, στα πλαίσια του πολιετούς ε, δημοσιονομικού ε, πλαισίου 2014-2020 και χαίρομαι ιδιαίτερα και για τις τεράστιες αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο κόσμο που συνεχώς ενεξελίξει. Θα διευκολυνθούν έτσι οι τρόποι χρηματοδότησης, οι διαδικασίες και θα τίνουμε προς, ε, στόχους, προς τους στόχους της στρατηγικής 2020. Ε, Εγώ συγχαίρω τον κύριο Σιμάνσκι για την εργασία του και τις προτεραιότητες που δίνει στον τομέα της ενέργειας. Να τίνουμε προς μια κοινή αγορά εξωτερική αγορά για την ενέργεια και αυτό φυσικά χρειάζεται την άμεση συνεργασία με τους εταίρους μας. Η μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών μέσων για την ευρωπαϊκή πολιτική γυτνίαση βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες, τη διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες, την διασυνοριακή συνοχή και την ευελιξία των προγραμμάτων. Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες ε, γύρω από τις οποίες εγώ θα βασίσω τις θέσεις μου. Θα εισάγω και τις σχετικές ε, τροπολογίες σε όλους τους, για όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας και πιο συγκεκριμένα την υποστήριξη των ΜΜΕ στην βιομηχανία, στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στις τηλεπικοινωνίες. Οι ανάγκες ε, των χωρών εταίρων πρέπει να οριστούν. Πρέπει να ορίσουμε τις ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές, να ορθολιγοποιήσουμε τα προγράμματα για να έχουμε πιο αποτελεσματική και πιο, πιο αποτελεσματική βοήθεια. Ε, γιατί η επιτυχία χρειάζεται και διάρκεια. Είναι σημαντικές οι προκλήσεις για το μέλλον, συνολικά για όλο τον πλανήτη. Μπορούμε εμείς με όλα αυτά τα δημοσιονομικά μέσα να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους σε όλα τα επίπεδα και να προτίσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και να διασπαλίσουμε και αηφόρο ανάπτυξη για τους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σιμάνσκι για τη δουλειά του. Ήδη ξεκινήσαμε τις συζητήσεις και θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η ασφάλεια τροφοδότησης σε ενέργεια αποτελεί το βασικό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό χρειάζεται καλή συνεργασία με τους γειτόνους. Συνεργασία που θα πρέπει να βασίζεται σε μια ρυθμιστική ολοκλήρωση των αγορών, διαφοροποίηση των πόρων και των διαμετακομιστικών οδών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ορίστηκε από το Συμβούλιο ε, όριο για την ε, ολοκλήρωση της ε, κοινής αγοράς ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καλό θα ήταν να προσυπογράψουν οι γειτονέ μας την συνθήκη ε, και το πρωτόκολλο για την ενέργεια, όπως επίσης και για τους τρόπους διαμετακόμισης. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συμπληρωματικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ολοκλήρωση ε, των περιφερειακών πολιτικών με τις στρατηγικές του 2020 θα καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες για την ενίσχυση της ενεργειακής πλευράς της πολιτικής γυτνίασης με τις χώρες του Νότου και τις άλλες όχθης της Μεσογείου λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Ευχαριστώ η συνάδελφος Μπαλεάνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ την εισηγητή γιατί νομίζω ότι η εργασία του είναι πολύ ολοκληρωμένη και ισορροπημένη. Αυτά που είπατε κύριε Σιμάνσκι για την εσωτερική αγορά ενεργείας είναι κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα. Υπάρχουν όμως και ορισμένα θέματα που θέλω να σχολιάσω. Πρώτον φοβάμαι ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνουμε στα λόγια διότι συνεχώς λέμε στους γείτονές μας πόσο σημαντικοί εταίροι είναι ενεργειακός αλλά γνωρίζουν πολύ καλά, α, το ξέρουν ήδη πολύ καλά και γι' αυτό οι ανατολικοί μας γείτονες παίρνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Μερικοί από αυτούς είναι πολύ δυναμικότεροι από μας από και από ό,τι πιστεύουμε για εκείνους. Δεύτερον, για να δημιουργηθεί μια πραγματική αγορά, εσωτερική αγορά του αερίου, πρέπει να εξισορροπηθούν και οι δύο πλευρές και η αλληλεξάρτηση. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε κοινά πρότυπα με βάση τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, αλλά εδώ παίζεται η αξιοπιστία μας. Πώς να ζητήσουμε από τους εταίρους μας να απελευθερώσουν τις αγορές τους όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει καν τη δική μας. Έχουν γίνει πολλές προσφυγές καταχωρών για μη εφαρμογή της ενεργειακής δέσμης. Τέλος, Έχουμε πολλά εργαλεία για τη διεθνή συνεργασία με βάση μεταξύ άλλων και την ενεργειακή χάρτα αλλά πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε με τους εταίρους μας για τα ενεργειακά, αν θα υπάρξει ο προτινόμενος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών και αυτά που συζητάμε σήμερα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα νομοθετήματα θα συμφωνούν μεταξύ τους και το μήνυμά μας να είναι συνεπές και απλό. ώστε να υπάρχει αμοιβαίο όφελος, συνεργασία κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Τελευταία η κυρία Ριβάζη. Ορίστε. Ριβάζη. Έφυγε Ριβάζει, ριβάζει. Όχι. Τότε ο εισηγητής. Ε, η τωρινή κατάσταση είναι προσωρινή. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν χρειαζόμαστε μία συνεπή θέση και άρα να ενδυναμωθεί η έκθεση με συμπερίληψη και των θεμάτων ενέργειας και συνεργασίας. Let's do it. Ευχαριστούμε. Let's do it. Ζητώ συγγνώμη από τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών για την καθυστέρηση Τετάρτη στις 12 λίγη διορία κατάθεση τροπολογιών και η επόμενη μας είναι